Λοιπόν, οι αρμόδιες αρχές της ε, Ρουμανίας μου μετέφεραν την αντικατάσταση της κυρίας Κρέτου από τον κύριο Πάβελ από τον Νοέμβριο του 2014 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης που διέπει την εκλογή ε, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρθρο 4 παράγραφη 1 και 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την ε, ε, εκλογή του κυρίου Μίλαν Πάβελ. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, εφόσον δεν έχουν ακόμα επαληθευθεί τα διαπιστευτήριά του, ο κύριος Πάβελ θα συνεχίσει να συμμετέχει στα όργανα και στις εργασίες έχοντας υπογράψει επίσης και την δήλωση ότι δεν είναι πλέον, ότι μπορεί να συνεχίσει να είναι ε, βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και μια αντιπροσωπεία της Καναδικής Βουλής Προεδρεύεται η αντιπροσωπεία του Καναδά. Προεδρεύεται